έχουμε το θέμα της ε, αντίθεσης για το Λουφοζάτ. Ο κύριος Λαβία, τέσσερα λεπτά. Grazie Presidente, signor Commissario, colleghi. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή συζήτηση δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα ύψης της σημασίας που αφορά την ανθρώπινη υγεία, την αγία των ζώων και το περιβάλλον. Χαίρομαι λοιπόν, διότι η συζήτηση αυτή βρίσκεται ενώπιον όλων. Είχαμε πολλές συζητήσεις σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανανέωσης της χρήσης του γλυκοσέιτ Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ε, φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η ουσία αυτή είναι μια δραστική ουσία που στην ουσία ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να μολύνει το περιβάλλον παγκόσμια. Χρησιμοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά το 76% χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό και θίξαμε αυτή την αντίρρηση ζητώντας από την Επιτροπή να αποσύρει το κανονισμό εκτέλεσης έτσι ώστε να έχουμε ένα σαφή κατάλογο νέων ή παλαιών νησιών που δεν μπορούν να τεθούν σε εμπορία. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μία αναθεώρηση της ταξινόμησης του γλυφοσάτ με βάση τα προϊόντα που είναι ε, διαθέσιμα και το γεγονός ότι αυτή η δραστική ουσία μπορεί να προκαλέσει και καρκίνο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτό το δεδομένο που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Το Μάρτιο του 2015 ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας με τον, για τον καρκίνο θεώρησε το γλυφοσάτ ε, ο, θεώρησε το γλυφοσάτ προκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο και είχε επαρκή στοιχεία για να μιλήσει και για νεοπλασίες στα ζώα. Το 2015 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, προέβη μία αξιολόγηση του γλυφοσάτ και έκρινε ότι μάλλον αυτό το προϊόν δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο και γι' αυτό δεν θα πρέπει να ταξινομηθεί ε, ως προκαλών καρκίνο. Και γι' αυτό μέσα στα πλαίσια των ε, φυτοφαρμάκων έκρινε ότι θα μπορούσε αυτό το προϊόν να τεθεί σε εμπορία. Θα πρέπει όμως να ακολουθήσουμε μία προληπτική οδό έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να μην έχουν ε, αρνητική επίπτωση στον άνθρωπο και στα ζώα. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να τηρήσουν την αρχή της πρόληψης όταν στον επιστημονικό τομέα υπάρχουν ε, στοιχεία που δεν είναι απόλυτα σαφή σε σχέση με την ε, ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό η Επιτροπή Περιβάλλοντος θεωρεί ότι ο κανονισμός ε, δεν ε, τηρεί την αρχή της πρόληψης και δεν, δεν τηρεί το κανονιστικό πλαίσιο. Ζητούμε από την Επιτροπή να αποσύρει αυτό το σχέδιο κανονισμού και ζητούμε από την ΕΦΣΑ να μας δώσει όλα τα επιστημονικά στοιχεία. Πρέπει να, να ολοκληρώσετε. Εξ ονόματος βεβαίως της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την οποία και εκπροσωπώ. Μερος Επιτροπής, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω πως το δικαίωμα ε, επαλήθευση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά το γεγονός κατά πόσον η υλοποίηση του κανονισμού ξεπερνά τις, ε, το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το κανονιστικό κείμενο. Η εφαρμοστική λοιπόν πράξη σχετική με το γλυφοσάτ στηρίζεται στο κείμενο του κανονισμού 1107 του 2001 και 1982 του 2011 για την επιτροπολογία. Η Επιτροπή θεωρεί ως εκ τούτου πως δεν, δεν υπερεύει τις εφαρμοστικές της εξουσίες. Έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο εφαρμοστικής πράξης στην μόνιμη υποεπιτροπή σε σχέση με το ε, νομικό πλαίσιο. Οι υπηρεσίε Επιτροπής αυτή τη στιγμή συνομιλούν με τα κράτη-μέλη για να προσδορίσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανανέωση της ε, υλοποίησης της διάταξης σχετικά με το γλυφοσάτ με την ε, μέγιστη δυνατή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Το σχέδιο εφαρμοστικής πράξης εκ τούτου θα τροποποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα και δεν μπορεί να θεωρείται ως απόφαση της Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, πριν τοποθετηθείτε για το σχέδιο ψηφίσματος, θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία ήδη ε, είχαν επισημανθεί κατά την ε, συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου. Το σχέδιο κανονισμού καταγράφει μια ρητή δέσμευση σχετική με την ανανέωση της άδεια, εάν έχουμε στοιχεία ταξινόμη σχετικά με την ε, έγκριση. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο με στοιχεία που δεν θα επέτρεπαν το τα προϊόντα που περιέχουν γλυφοσάτ να διατίθεται στην αγορά εφόσον υπάρχει το τελοουάμιν που θεωρείται co-formulant. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τον κλάδο, το παραγωγικό, να δημοσιεύσει τις σχετικές μελέτες και θα ήθελα ιδιαίτερα να παραπέμψω στι εργασίε τη Task Force τη σχετική με τον γλυφοσάτ. Έχουμε λάβει τι σχετικέ ε, απαντήσει και τώρα διευκρινίζουμε τι λεπτομέρειε του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τώρα, 1,5 λεπτό, η κυρία Ντελάη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα Πρόκειται για μία ένσταση σε ό,τι αφορά την εκτελεστική πράξη, και έτσι δεν έχει καμία νομική προέκταση. Όμω, συμμερίζομαι τι ανησυχίε ορισμένων πολιτών και παράλληλα υπάρχει και μία ανεφρεγουμένου κρίση στο γεωργικό κόσμο. Πολλοί γεωργοί χρησιμοποιούν στην Ευρώπη το γλυφοσάντ. Είναι θεμελιώδη σημασία λοιπόν αυτή η ουσία ω ζενιοκτόνο. Δεν υπάρχει ε, άλλη βιώσιμη εναλλακτική που να προτείνεται στους γεωργούς. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει ε, αυτό το, αυτή η στενοπός που, στην οποία έχουμε βρεθεί τώρα να ε, επιληθεί. Και εμεί έχουμε ψηφίσει επί του ζητήματο στο παρελθόν και έχει τηρηθεί και η διαδικασία. Επιπλέον, σε περίπτωση νέων στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα μπορεί να αναθεωρήσει την ε, άδεια που έχει δώσει. Και σίγουρα μέχρι το 2017. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει τροπολογίες εκ μέρους ε, ε, του ΕΛΚ ε, θέτοντα ορισμένου περιορισμού, ζητώντα την επιτάχυνση του καταλόγου των βοηθητικών ουσιών που θα πρέπει να απαγορευτούν, όπω η τελαβαμίνη, και ε, θέτουμε και ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για τα κράτη-μέλη. Να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε την έρευνα και κοινοτομία για να βρούμε εναλλακτικέ λύσει προ το γλυφοσάτ. Και ε, συνιστώ σε όλου του συναδέλφου να στηρίξουν την πρότασή μου. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ την Πρόεδρο, την συναδελφό. Έχετε μια μπλε κάρτα της κυρίας Μίλιος. Τη δέχεστε? Τη δέχεστε? Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δείξατε κάποια σημεία που έχουν να κάνουν με το γλυφοζάτ και τη χρήση του. Δεν ε, αναφερθήκατε όμως στο γεγονός ότι εισάγουμε κτηνοτροφές από τρίτα κράτη, γιατί και αυτό είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί εν προκειμένου. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εάν με βάση την αρχή της πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρούσατε ότι θα έπρεπε να ταχθούμε κατά το περαιτέρω χρήσης γλουφοζάτ ε, και σε τρόφιμα και σε ζωοτροφές. j'espère avoir compris euh, d'après la, transcription. Ευχαριστώ. Ε, από τα όσα κατάλαβα την ερώτηση σας, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όντως συζήτηση ευρύτερη στην υπόθεση αυτή πριν να καταλήξουμε σε μια οριστική απόφαση. Ο Πρόεδρος, εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Πότς, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το πιο θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να διατυπώσει αντιρρήσει κατά εκτελεστικών εφαρμοστικών πράξεων τη επιτροπή. Είναι το θλιβερότερο στοιχείο αυτό και αποκαλύπτει τις αδυναμίες τη διαδικασία ε, της Επιτροπολογίας. Αυτό ρίχνει όλο και πιο δυσμενές φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν αφήνει κατάλοιπα το γλυφοσάτ στις ΗΠΑ. Γίνονται τώρα έλεγχοι παρουσίας γλυφοσάτ στα τρόφιμα και πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουμε το καταναλωτή. Η ΕΦΣΑ ε, αιτιολογεί και στηρίζει τις αποφάσεις σε κάποιες μελέτες οι οποίε όμως είναι μυστικέ και τι οποίες έχει χρηματοδοτήσει ο παραγωγικός κλάδος. Πάντω φαίνεται ότι το γλυφοσάτ έχει χαρακτηριστεί υπεύθυνο για πολλές ασθένειες, πιθανώ υπεύθυνο για πολλέ ασθένειε και ε, διαταράξει του ενδοκρινικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκέρλινγκ, ECR. Ε, μισή λεπτό. Thank you very Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου θα αντιταχθεί στεναρά σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Θα μπορούσα να σας ε, μιλήσω επί μακρόν για τη χρήση του γλυφοσάτ και πόσο μεγάλη σημασία έχει στη γεωργία. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για τις ελλείψεις του ψηφίσματος. Το ψήφισμα ορίζει και λέει ότι βρεθήκαναν υπολείμματα γλυφοσάτ στη γη και στον υδροφόρο ορίζοντα. Αλλά όπως μας λέει και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Κινδύνων, ε, μας μιλά για ένα 1% ή κάτω από το 1% υπολείμματων. Επίσης υπάρχουν υπολείμματα στα τρόφιμα. Δεν πρόκειται για κινδύνους όμως, για πραγματικό κίνδυνο και έχουμε να κάνουμε με επίπεδα πολύ κατώτερα και δεν πλήττουν την ανθρώπινη υγεία. Γιατί λοιπόν προβάλλεται αυτή η στάση η οποία δεν έχει και σημασία επί της ουσίας. Στο J αναφέρεται ότι τρέχουν σαν πρόταση δεν έχει περιορισμού στη χρήση. Αυτό δεν ισχύει γιατί ο κανονισμός εφαρμογής ορίζει ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με τη χρήση των δραστικών αυτών ουσιών. Άρα, πριν καν σκεφτούμε για τη χρήση του γλυφοσάτ και ε, την αξία που έχει, θα πρέπει να είμαστε σαφείς και όταν μιλάμε για την ε, αρχή της πρόληψης, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα πρέπει να καλύψουμε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη. Εδώ υπάρχει πληθώρα αποδείξεων και θα πρέπει να ε, επιλέξουμε μεταξύ της IARC και της EFSA. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να μετακινηθούμε από την EFSA. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό. Άλντε Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς που είδα πότε θα γίνει η δημόσια συζήτηση στην Ολομέλεια, γιατί κατά τύχη είδα ότι γίνεται τώρα. Είναι δύσκολη όλη η διαδικασία της αδειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, τι είδους διαδικασία είναι αυτή όταν η Επίτροπος μετά την αδειοδότηση στέλνει επιστολές στο μεγαλύτερο βιομηχανικό γίγαντα του κλάδου, ζητώντας περισσότερη διαφάνεια. Υπήρξαν λοιπόν τεράστιες δυσκολίες και όντω έχουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή την ΕΦΣΑ, έχουμε την ε, διαδικασία της αδειοδότησης και η ΕΦΣΑ είναι ξεκάθαρη στη δήλωσή της. Η ομάδα μου λοιπόν θεωρεί ότι θα πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή τα όσα λέει η ΕΦΣΑ. Δεν αναφέρει λοιπόν τίποτα για τον χρονικό ορίζοντα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γι' αυτό και έχουμε υποβάλει τροπολογία ως φιλελεύθεροι, με την οποία καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει την αδειοδότηση του γλυφοσάτ αλλά για μια περίοδο 5 ετών κατά μέγιστο και να λάβει υπόψη τυχόν νέα στοιχεία μέχρι τότε που θα αποδεικνύουν ότι αυτή η ουσία είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι νομίζαμε και θα πρέπει να αποσυρθεί η αδειοδότηση. Αυτή είναι η τροπολογία που υποβάλαμε πριν από 20 μόλις λεπτά και ελπίζω να μπορέσετε να την στηρίξετε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη προς τους συναδέλφους ε, Γκέρλινγκ και Σάνι. Υπήρχε μπλε κάρτα για σας κυρία Γκέρλινγκ. Θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ κύριε Σάνι αν θέλετε να αποβάλλετε το ερώτημά σα, Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γκέρινγκ κάτι το οποίο εντάσσεται στην όλη συζήτηση. Εάν υπάρχει τέτοια αντίσταση στην χρήση ε, του γλυφοσάτ, παρότι έχουμε τεράστια χρήση, 50% ε, χρήσης ε, τέτοιων προϊόντων από αυτή τη βιομηχανία. Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστώ, αν κατάλαβα καλά. Ρωτάτε για την χρήση του λιφοσάτ. Μιλήσατε για κακάο, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι σας κατάλαβα καλά. Είναι πολλές οι ε, και οι γεωργικές εφαρμογές ε, και σε τελευταία ανάλυση πολλέ είναι πολύ πιο σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτήν τη παραγωγής ε, κακάο. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, η χρήση, είναι σημαντική, γι' αυτό υπάρχει και η οδηγία για την ε, αηφορία στην γεωργία που δίνει οδηγίες προς τους γεωργούς ως προς τη χρήση και τους όρους χρήσης του γλυφοσάτ και μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση προβλημάτων. Βεβαίως και μπορεί να αντιμετωπιστεί αντίσταση, αλλά νομίζω ότι όντως χρειαζόμαστε το γλυφοσάτ. Ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος της ε, ΓΟΕ, η κυρία Κιούλορεν. Ένα λεπτό. Πρόεδρε. Το γλυφοζάτ. Το Μάρτιο του 2015 χαρακτηρίστηκε από την ΕΑΣΥ ε, καρκινογόνος ουσία. Άλλωστε υπάρχουν και στοιχεία πως πρόκειται για ενδοκρινικό διαταράκτη. Μάλιστα με βάση κάποια στοιχεία χρειάζεται δύο εβδομάδες λένε για να ε, εξαφανιστεί η δράση του από το περιβάλλον αλλά αυτό δεν αληθεύει διότι υπάρχουν και άλλα παράγωγά του όπως το ANPVA ε, ε, που περνούν στο έδαφος και δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ιδιαίτερα σε ψυχρά κλίμακα, κλίματα. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη λοιπόν όταν γίνονται μελέτες, γιατί οι μελέτες αυτές έλαβαν χώρα σε ε, περιοχές με πιο θερμό κλίμα και διαφορετικούς τύπους ε, εδάφους. Πρέπει να δούμε σε περιοχές με πιο ψυχρό κλίμα πώς ε, γίνεται η, ποια είναι, ποιος είναι ο κύκλος ζωής του γλυφοσάτ. Και τώρα ο Μάρτιν Χόιστιν λέει μέρος των πρασίνων, 1,5 λεπτό. Ναι, χαίρομαι που συζητούμε το γλυφοζάτ αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, διότι Έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η αρχή της πρόληψης. Την ε, στον κίνδυνο για καρκίνους δεν τον ανέφερε κάποιος τυχαίος, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Και υπάρχουν πάρα πολλές ε, έρευνες από πανεπιστημιακά ιδρύματα που εξετάζουν την ε, κατάσταση αυτή που οδηγεί σε συμπεράσματα πως μέχρι και 70% αύξηση των ε, καρκίνων έχουμε συνδεόμενων με το γλυφοσάτ, ε, το οποίο είναι παρόν σε άπειρα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και η μπύρα και πολλά άλλα. Κυρία Γκέρλινγκ, πρέπει να κοιτάξουμε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να σκεφτούμε με σοβαρότητα, καταρχάς αν υπάρχουν εναλλακτικέ και δεύτερον, εάν είναι δυνατόν να δεχθούμε μετά από μια διαδικασία μακροσκελής συζητήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χωρίς κανένα περιορισμό ανανεώνεται η άδεια για 15 χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι δεν γίνεται καμία έρευνα, δεν γίνεται καμία μελέτη και μόνο με όρους οικονομικούς, γιατί κερδίζει, ε, εξοικονομεί χρήματα ο Γεωργός, ε, θα χρησιμοποιείται και πάλι το γλυφοζάτ, χωρίς να υπάρχουν ε, μελήματα ούτε οικολογικού, ούτε, σχετικά, ούτε οικολογικού χαρακτήρα, ούτε σχετικά με τη δημόσια υγεία. Χρειάζεται να εξεταστεί με μεγαλύτερη διαφάνεια, με βάση και την λεγόμενη αρχή της διαφάνειας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπάρξει διαφάνεια γενικότερη και όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λύση έχει μια μπλε κάρτα για σας αν τη δέχεστε. Μάλιστα. Παρακαλώ κύριε Λύση. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χόισλινγκ. Είπατε εσεί ότι δεν έχει προτείνει περιορισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, στι τροπολογίε όπω αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο γίνεται λόγο για περιορισμού, όπω ακριβώ του ε, ζητάτε κι εσεί και μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ ε, πιο προσεκτικά τα αιτήματα αυτά, εάν δηλαδή υπάρξουν περαιτέρω στοιχεία, θα κατατασσόταν το γλυφοζάτ σε, ε, επικίν, στις επικίνδυνες ουσίες και θα μπορούσε και να απαγορευτεί ακόμα. Δεν σας καλύπτει αυτό ως πράσινο. Κύριο Χόισλινγκ, χαίρομαι που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αυτό το μεγάλο άλμα προ τα μπρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα στην προστασία τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε τη βασική αρχή ότι δεν υπάρχουν απλώ χημικέ εναλλακτικέ στο γλυφοζάτι. Γιατί το πρόβλημα γλυφοζάτι, η χρήση του, είναι ότι υπάρχουν μηχανισμοί ε, που μπορούν με μηχανικά μέσα να αντικαταστήσουν έως και 90% τη χρήση του γλυφοζάτ. Γι' αυτό λοιπόν το κατά πόσον θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε απεριόριστα τέτοιου είδου ουσίε είναι ε, ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να κρυθεί μόνο με βάση την αρχή τη πρόληψη, Ο πρόεδρο. κοιτάξτε, κανονικά επιτρέπω μόνο μία μπλε κάρτα, αφήνω μόνο μία μπλε κάρτα να ομιλητεί, αλλά βλέπω και την κυρία Ιούσο. Αν τη δέχεστε, να την επιτρέψω. Κυρία Ιούσο. Μπορείτε να μου πείτε πόσο στοιχίζουν αυτά τα μέτρα και πόσες επιπτώσεις θα έχουν στο, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι επιπτώσεις θα έχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κύριος Χόισλινγκ, να σας πω. Εγώ έχω μια βιολογική γεωργική εκμετάλλευση και δεν χρησιμοποιούμε γλυφοσάτα εδώ και 30 χρόνια. Σας παρακαλώ να έρθετε να δείτε πώς λειτουργεί. Είναι απόλυτα εφικτό και αποτελεί μια ε, απόλυτη εναλλακτική. Ο πρόεδρο, κυρία Γκέρλινγκ, δεν μπορώ να σα επιτρέψω μπλε κάρτα γιατί είσαι στον κατάλογο των ομιλητών. Παρακαλώ και εσεί να δείξετε κατανόηση. Τώρα εκ μέρου τη EFDD, η κυρία Εύη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση επειδή ακριβώς ε, θα ψηφίσουμε την Τετάρτη η αναθεώρηση του πλαισίου, μάλλον η ανανέωση της άδειας θα πρέπει να ανατραπεί. Δεν μπορούμε να ε, χρηματοδοτούμε μεγάλους κολοσσούς και τη στιγμή που δύο μεγάλοι οργανισμοί διαφωνούν θα πρέπει να μην ανανεωθεί η αδειοδότηση του προϊόντος. Όπως είπαμε υπάρχουν πολύ πολλές επιπτώσεις σε σχέση με ενδοκρινικές διαταραχές και γι' αυτό ακριβώς τους επόμενους μήνες θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση διεθνών οργανισμών. Πριν δεν θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε την άδεια. Επίσης υπάρχουν επιπτώσεις και στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό, κυρία Μαγκίνες. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η αλληλογραφία που έλαβα για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένα ευρύτατο λόμπι για την απαγόρευση του γλυφοσάτ και σεβόμαστε και όσους μας έστειλαν mail για αυτό το αντικείμενο. Όμως προσφάτως λαμβάνω και mail από μεμονωμένους Γιώργους και το χαιρετίζω αυτό, όχι από γεωργικές ε, αλλά από μεμονωμένου γεωργού που λένε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά την βιολογική γεωργία και την προσπάθεια περιορισμού του ε, οικολογικού αποτυπώματος ε, του γεωργού με έναν θετικό προς το περιβάλλον τρόπο. Είναι εύκολο να πει κανεί ότι πρέπει να απαγορευτούν τα χημικά. Ε, Όμω πρέπει να εξετάσουμε ακριβώ περί τίνο πρόκειται. Από ό,τι φαίνεται έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές επιστημονικές αξιολογήσεις, όμως μία, η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, εξετάζει τους κινδύνους, ενώ ο άλλος οργανισμός για τον καρκίνο εξετάζει τα ρίσκα, τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Νομίζω ότι είναι πολύ μετρημένη η θέση του Λαϊκού Κόμματο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ασφαλή τα προϊόντα, όμω δεν θέλουμε και πλήρη απαγόρευση. Στηρίζουμε την επαναδιοδότηση του προϊόντος, αλλά όχι για 15 χρόνια και θέλουμε να λάβουμε υπόψη τυχόν στοιχεία στο μέλλον. Να ακούσουμε λοιπόν όλες ε, τις φωνές ε, που ασκούν πιέσεις για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Η κυρία Κατενμπάχ. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, μιλούμε για το γλυφοσάτ, το οποίο χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή φυτοπροστατευτικό προϊόν, αλλά δεν είναι φυτοπροστατευτικό προϊόν, είναι ζυζανιοκτόνο. Φωνεύει τα φυτά και δεν κάνει διακρίση, ούτε κάνει ζυζανιοκτόνο μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, γιατί δεν κάνει διάκριση μεταξύ ζυζανίου και ε, υγιούς ε, φυτού. και φαίνεται ότι έχει κάνει η Μονσάντο μια προσαρμογή γενετική με ένα ένζυμο το οποίο επιτρέπει να είναι και ανθεκτικό το φυτό στο γλυφοσάτ το, οποίο είναι σε θέση να προξενήσει σημαντικές ε, ζημίες στον ανθρώπινο οργανισμό, διαταραχή των, της ενδοκρινικής λειτουργίας και των ορμονών. Άρα το θέμα είναι εάν είμαστε εκτεθειμένοι σε κίνδυνο. Δεν μπορούμε να αρνούμεθα ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά με το κλειφοζάτ. Εάν δεν υπήρχαν θα μπορούσαμε να το εγκρίνουμε, να δεχθούμε την αδειοδότηση. Αλλά αν λέμε ότι και κίνδυνος υπάρχει και δυναμικό ε, ζημίας, τότε δεν είναι δυνατόν να ανανεωθεί ή να παραταθεί η άδεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόκοβιτς έχει μια μπλε κάρτα για σας, κυρία Κάτινμπαχ. Τη δέχεστε. Με ακούτε κυρία Μπακάντμπαχ. Να τη δώσω. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφο το εξής. Εγώ ασχολήθηκα με τα οποροφόρα από το 86 και χρησιμοποιούσα το γλυφοσάτ ως ε, ζυζανιακτόνο για τα υποροφόρα και πολλοί από εμά ε, όταν το χρησιμοποιούμε θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η απόλυτη αλήθεια. Ιδιαίτερα γνωρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί για 40 χρόνια και κατά τη χρήση αυτή, μάλλον η χρήση αυτή δεν μας δείχνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον προληπτικό αποκλειστικά κίνδυνο. Κύριε Μπογκοβίτ, ε, βάλτε τα ακουστικά σα παρακαλώ. Κοιτάξτε, το νόημα τη μπλε κάρτα είναι να κάνετε ερώτηση στον ομιλούντα, όχι να αξιοποιήσετε το χρόνο για να κάνετε δηλώσει. Κυρία Κάτιντραχ, νομίζω δεν ε, υπάρχει λόγο να δώσετε απαντήσει και συνεχίζω τον κατάλογο των ομιλητών με την κυρία Σαλτμόζε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ μας ενδιαφέρει ε, η ταξινόμηση σε σχέση με τον ε, κίνδυνο ως προς τον καρκίνο. Υπάρχει μια τέτοια ε, πιθανότητα, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο ένας μεγάλος οργανισμός λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου. Μιλάμε λοιπόν για δύο διαφορετικές αξιολογήσεις. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να μας απασχολήσει γιατί αν γίνει αυτή η αδειοδότηση για τα επόμενα 15 χρόνια, τη στιγμή που υπάρχουν δύο διαφορετικές γνωμοδοτήσεις, θα έπρεπε να είμαστε απολύτως σίγουροι. Γιατί η ανθρώπινη υγεία θα πρέπει να προτάσεται του χρήματος. Θα πρέπει να εξεταστεί πλήρως το γλυφοσάτ πριν γίνει η νέα αδειοδότηση για τα επόμενα 15 χρόνια. Ίσως είναι δύσκολο να βρούμε εναλλακτικέ ουσίες, εναλλακτικά οκτώνα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε υπόψη των ΠΟΗ. Ευχαριστώ. Περνάμε στη δικασία Καρστιάη και πρέπει να σας ενημερώσω πως έχω αρκετά αιτήματα καθώς δεν είχα επαρκή χρόνο δεν μπορώ να τα μετρήσω, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να δείξετε και κατανόηση για να αφήσουμε και το χρόνο για, τις επόμενες, για τα επόμενα θέματα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είμαι επεπισμένη πως πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τι ψηφίζουμε εδώ. και να κρίνουν το θέμα της αδειοδότησης χημικών που χρησιμοποιούνται στην γεωργία και αν αυτά έχουν επίδραση στην ανθρωπινή υγεία. Καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να κρίνει κατά προτεραιότητα και να αποφασίσει τα θέματα αυτά. Έχω επικοινωνήσει με το τσεχικό Υπουργείο Γεωργίας και, ε, και το Υπουργείο Προστασίας του Καταναλώτη, τα οποία έχουν συμμετάσχει στη δικασία αυτή της αδειοδότησης και μου έχουν δηλώσει πως θα υποστηρίξουν την Επιτροπή στην αποφασή της. Θα υποστηρίξω λοιπόν και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί όπου γίνεται λόγος για περιορισμό της ε, χρονικής διάρκειας στα 7 χρόνια για την αδειοδότηση. Ευχαριστώ. Η επόμενη μελήτρια. Ευχαριστώ, λέει κυρία Γκαρσία. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί υπάρχουν αμφιβολίες που θα πρέπει να διασαφινιστούν. Είναι πολύ σοβαρό το ότι μερικοί συνάδελφοι λένε ότι υπάρχουν διαφορετικοί οργανισμοί με διαφορετικές γνωμοδοτήσεις. Όχι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σε σχέση με τη δραστική ουσία. Επίσης, το, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός από τη Γερμανία για την αποτίμηση, αποτίμηση κινδύνου μας λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ως προς το τελικό ζυζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται. Φυσικά είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιούν οι γεωργοί ευρέως, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΦΣΑ ή όχι. Εγώ προτιμώ να δείξουμε εμπιστοσύνη στο δικό μας ε, όργανο απόφασης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ashworth, για ένα λεπτό. Uh, Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο όμως θα πρέπει να είναι διασφαλίσει ότι τα ε, τρόφιμα είναι ασφαλή και υπάρχει και χρηστή διαχείριση του περιβάλλοντο. Και αυτή είναι μια πολύ ε, σημαντική ευθύνη την οποία πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά. Από την άλλη, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι αποφάσει που λαμβάνουμε είναι αυστηρά αναλογικέ ω προ ε, τον κίνδυνο και όχι την έκθεση σε κίνδυνο, το hazard. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τι συνέπειε αυτών των αποφάσεων. Στην περίπτωση που ένα προϊόν το οποίο έχει υιοθετήσει και εγκρίνει αν θέλετε η ΕΦΣΑ και δεν υπάρχει και ένα άλλο εναλλακτικό προϊόν, ε, για να το αντικαταστήσουμε κάτι άλλο, η βιομηχανή θα πρέπει να επανέλθει σε πιο παραδοσιακές ε, μεθόδους και θα πρέπει να επανέλθει σε αύξηση της χρήσης άλλων ε, αγροχημικών προϊόντων και αυτό θα έχει πολύ σημαντικές προεκτάσεις ε, για μια βιομηχανία που ήδη δέχεται μεγάλες πιέσεις. Πρέπει λοιπόν να μας ε, διακατέχει περισσότερο η λογική και όχι το συνέστημα. Γι' αυτό θα πρέπει να το υιοθετήσουμε. Κυρία Πίτερ. Ευχαριστώ. Το Διεθνές ε, Ερευνητικό Κέντρο για τον Καρκίνο έχει αναφέρει ότι ενδεχομένως να είναι καρκινογόνος ουσία το γλυσοφάτ. Σε διάφορες μελέτες βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ε, πρόκλησης ε, λεμφώματος σε όσους έρχονται σε επαφή με το γλυφοσάτ. Βεβαίω, οι εταιρείε δεν μα το λένε αυτό γιατί θέλουν να απολύσουν γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού που θα είναι συμβατοί μόνο με το γλυφοσάτ. Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση για την επιμήκυνση τη αδειοδότηση ε, ε, του γλυφοσάτ μπορεί να γίνει μόνο με την τήρηση της αρχής της ε, αναλογικότητας, μάλλον της προφύλαξη οι εμπειρογνώμονες λένε ότι ο αντίκτυπος ε, του γλυφοσάτ ε, στην ανθρώπινη υγεία ε, φαίνεται μέσα στον πρώτο χρόνο και έχοντας κατά νου και το εύρος των επιπτώσεων για την υγεία. Ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι διατηθμένη να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το γλυφοσάτ. Γι' αυτό θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμπεριφέρεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτε και μάλιστα φαίνεται και να λησμονεί να λησμονεί σκάνδαλα σοβαρά όπως αυτό το σχετικό με την γερμανική μπύρα και δεν λαμβάνει υπόψη προειδοποιήσεις των ερευνητών που λένε ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία το γλυφοσάτ. Μπορεί να είναι ίσως πρόημο το να ζητήσει κανείς απόλυτο, απόλυτη απαγόρευση του κλειφοσάτ σε μια εποχή όπου η γεωργία βρίσκεται σε κρίση και αν απαγορεύσει το κλειφοσάτ θα βρεθεί σε ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία ο Ευρωπαίος Γεωργός. Γι' αυτό θεωρώ ότι το καλύτερο σήμερα θα ήταν να δοθεί παράταση στην άδεια του κλειφοσάτ για ένα-δύο χρόνια το πολύ αλλά να καταστούν και πιο αυστηροί κανόνες σχετικοί με την χρήση του. Θα μπορούσε παραδείγματι να απαγορευτεί η χρήση του στην περίοδο που προηγείται τη συγκομιδής και να αναστηθούν βεβαίω εντωμεταξύ εναλλακτικέ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Ροπέ και έτσι ολοκληρώνεται τη διαδικασία Καριστιά εκ μέρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει στις πολυάριθμε ερωτήσει, κυρία Γιώρουβα. Αγαπητέ Πρόεδρε, μέλη, θα ήθελα να επαναλάβω ότι το επίδικο ζήτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοστεί μία κανονιστική ρύθμιση μέσα στα πλαίσια της βασικής αυτής πράξης. Όπως σας είπα, η απόφαση αυτή είναι συνεπής με το σχετικό κανονισμό γιατί, και γι' αυτό θεωρούμε ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες εκτέλεσης θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για την ανανέωση της χρήσης του γλυφοσάτ έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία των κρατών μελών. Άρα το, η, η νομοθετική πράξη, η πράξη κανονισμού θα τροποποιηθεί. Ο κύριος Τζοβάνι Λαβία έχει το λόγο, εισηγητής για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πολύ σημαντική γιατί μπορέσαμε ο καθένας να εκφράσει τη δική του θέση. Είδαμε ότι υπάρχουν διχογνωμίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως ε, ε, είχε προηγηθεί και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όμως υπάρχουν ε, λύσεις και μιλήσαμε για ορισμένες τροπολογίες πολιτικών ομάδων που θα μπορούσαν να μετριάσουν τις ε, απαιτήσει αυτές ε, ανανέωσης της άδεια, αλλά παράλληλα να έχουμε ένα πιο βραχυχρόνιο ορίζοντα για να δούμε κατά πόσο αυτό το προϊόν είναι καρκινογόνο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το προϊόν αυτό που χρησιμοποιείται ευρέως στη γεωργία χρησιμοποιείται ως ζυζανιοκτόνο και θα μπορούσε να αντικατασταθεί με μηχανικές ή χειρονακτικές εργασίες οι οποίες τεχνικώς είναι δυνατές όμως θα υπέσκαπταν την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού μας συστήματος. Γι' αυτό τις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε φυσικά και θα ήθελα να το σκεφτείτε. Ένα άλλο στοιχείο που ανέκυψε είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Τροφίμων. Είναι ο οργανισμός που έχουμε στη διάθεσή μας και όπως είπε και η συνάδελφος από τη σοσιαλιστική ομάδα, είναι το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη. Διαφορετικά, τι νόημα έχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που επιβαρύνουν και τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Λαβία. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση, κατατίθεται ψήφισμα, θα ψηφιστεί αύριο.